Κυρίε και κύριοι, μου ζητήθηκε να κάνω μια δήλωση για το τσουνάμι και την καταστροφή στη Φουκουσίμα. Και μετά τη δήλωσή μου θα ακολουθήσει συζήτηση με έναν γύρο από τον εκπρόσωπο της ε, κάθε ομάδες. Κυρίε και κύριοι, πριν από ένα έτος η Ιαπωνία επλήγει από μια τριπλή καταστροφή. Πρώτα απ' όλα υπήρχε ένα σεισμό της κλίμακας, 9 ε, βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κατόπιν ε, έπληξε ένα τσουνάμι ε, τμήμα της ακτής μήκους 400 χιλιόμετρων και μετά υπήρχαν εκρήξεις στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταΐτσι. Είχαμε μια τήξη του πυρήνα, τα χειρότερα γεγονότα από το Τσενομπίλ σήμερα τιμούμε τη μνήμη των 19.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, των χιλιάδων που έχασαν συγγενείς, τους 340.000 ανθρώπους οι οποίοι από την ακτινοπολία αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και όλους όσους έχασαν για πάντα το σπίτι τους. Το πώς αντέδρασε ο Ιαπωνικός λαός βεβαίως ήταν κάτι το οποίο συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο. Το θάρρος των ανώνυμων ηρώων στη Φουκουσίμα αυτών οι οποίοι πήγαν μέσα στον αντιδραστήρα και διακινδύνευσαν τις ζωές τους για να αποφύγουν τα χειρότερα ήταν κάτι το οποίο μας άγγιξε όλους. Η δύναμη με την οποία ο Ιαπωνικός λαός ρίχθηκε στο έργο της ανοικοδόμησης μας εντυπωσίασε όλους. Το Ιαπωνικό, το, ατύχημα στην Φουκουσίμα ξεκίνησε μια παγκόσμια συζήτηση για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, αυτή η συζήτηση γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο καθένας από εμά πρέπει να αποφασίσει μόνος του πού βρίσκεται όσον αφορά αυτή τη συζήτηση, αλλά είναι καλό το ότι λαμβάνει χώρα εδώ μέσα αυτή η συζήτηση, όσο επίμαχη και αν είναι, γιατί βεβαίως παρά το ότι το ενεργειακό μείγμα δηλαδή οι διάφορες πηγές ενέργειας και άρα η απόφαση υπέρ κατά της φυρνικής ενέργειας είναι εθνική αρμοδιότητα, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει κάθε κυβέρνηση και κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ευρωπαϊκή συζήτηση που πρέπει να γίνει γιατί στην Ευρώπη όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με τα δίκτυα ηλεκτρισμού του των γειτόνων μας. Το τι συμβαίνει σε μια χώρα επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων στις γειτονικές χώρες. Αυτή τη στιγμή 13% της ευρωπαϊκής ενέργειας παράγεται από την ελληνική ενέργεια και το εάν είναι αρκετά σίγουρη αυτή είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Βεβαίως η Φουκουσίμα είναι το χειρότερο ποινικό ατύχημα από την εποχή του Τσενομπίλ και ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Αυτό είναι το δίδαγμα το οποίο πρέπει να αντλήσουμε. Παρόλες τις διαφορές απόψεων μεταξύ όσων είναι υπέρ και κατά της ποινική ενέργειας, ένα είναι σαφές. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εγγυηθούμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτών. Σε αντίθεση με πολλούς που και μετά από αυτή την τραγωδία μόνο συζητούσαν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδρασε. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οπωσδήποτε των ειδικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν χώρα το έτος μας πέρασε για να γίνει πιο ασφαλής η πυρηνική ενέργεια. Σε αυτό ανήκουν σε αυτό λοιπόν, σε αυτές ανήκουν τα εθελοντικά στρες τεστ που έγιναν σε 143 πυρηνικά εργοστάσια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούνιο θα υποβάλει οριστική έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα εδώ πέρα να επαναλάβω την απέτησή μου. Όσα εργοστάσια δεν περάσουν αυτά τα stress test πρέπει να αποσυνδεθούν αμέσως από το δίκτυο και να τεθούν εκτός λειτουργίας. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται ένα τεστ, να μην περάσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο και να συνεχίσει να λειτουργεί. Χαιρετίζω επίση την έκθεση για τα πυρηνικά απόβλητα, την οποία εγκρίναμε πέρσι στο Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά υπάρχουν πανευρωπαϊκώς δεσμευτικοί κανόνες και προδιαγραφές για τα πυρηνικά απόβλητα. Επίσης ε, ψηφίστηκε το Φεβρουάριο μια έκθεση για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οικονομίες στις τάξεις του 20% για να έχουμε αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, κάτι το οποίο βεβαίω είναι ένα ορόσημο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας 2020. 20 Θα ήθελα λοιπόν από την καταστροφή στην Φουκουσίμα η οποία βεβαίως επέφερε τεράστιο πόνο να αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία πρέπει ανεξάρτητος του τι άποψη έχει ο καθένας υπέρ κατά της πυρηνικής ενέργειας είναι κύριο διδάγμα το ότι έχουμε μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας, ειδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα όπως το κάναμε και όπως πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το δίδαγμα και η προεδοποίηση της Φουκουσίμα είναι σαφές αυτό το οποίο είναι εφικτό δεν σημαίνει πως πρέπει οπωσδήποτε και να το πραγματοποιούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση επί των δηλώσεων του Πρόεδρου. Ο κύριος Οντί έχει τον λόγο για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Χθες στις 6.46 ώρα Στρασβούργου σταμάτησε, πάγωσε η ζωή στο, στην Ιαπωνία. Όλοι οι Ιαπωνέζοι σταμάτησαν τις ασχολίες τους έτσι ώστε να έχουν μια σκέψη, ένα λεπτό ε, στο οποίο να αναλογιστούν την καταστροφή που έγινε και τους ανθρώπους που υπέφεραν. Στις 11 ε, Μαρτίου ε, πριν από ένα χρόνο ένας σεισμός της τάξης των 9 βαθμών της κλίμακος Ρίχτερ δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα και σταμάτησε τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού. Δυστυχώς 55 λεπτά μετά κύματα ύψους 20 μέτρων ε, ε, οδήγησαν στην ε, ολική καταστροφή 340.000 εκτοπισμένοι, πολλοί νεκροί και την μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή του πλανήτη. Εξ ονόματος του ΕΛΚΑ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας και να πούμε ότι και εμείς έχουμε μια σκέψη για το κουράγιο και την αξιοπρέπεια των Ιαπώνων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Μετά από την καταστροφή αυτή ξεκίνησε, όπως υπενθυμίσατε, μια πολιτική συζήτηση ε, υπό το κράτος ε, του, συναισθήματο που προκλήθηκε από την καταστροφή, ορισμένες πολιτικές διοικήσεις πήραν κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Αλλά βεβαίως το, είναι σημαντικό το ότι το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας έχει τεθεί. Ε, προστίθεται δε εις ε, τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από τις φυσικές ε, καταστροφές, όπως ας πούμε του σεισμού της Αιτή. Ευχαριστούμε ε, κύρια ε, Επίτροπε γιατί και μετά από πρωτοβουλία του συναδέλφου σας ε, στις 24 και 25 Μαρτίου 2011 συνεκλήθη το Συμβούλιο έτσι ώστε να πάρει αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθη να αναθεωρήσει την οδηγία του 2009 ε, και επομένως ξεκίνησε μια διαδικασία ε, αναθεώρησης σε όλες τις χώρες. Το τέλος του 2012 θα έχουμε την πρώτη ενδιάμεση αξιολόγηση. Το ΕΛΚ επιθυμεί να ανοιχνευτούν νέες οδοί όσον αφορά πρώτον την ασφάλεια. Θα πρέπει να ε, εξασφαλιστεί ότι έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπέρ των πολιτών μας. Γνωρίζουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και επομένως θα πρέπει οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις και τα επιτεύγματα να επιβληθούν τους ε, εμπλεκόμενους φορείς θεωρούμε ότι βεβαίω ότι θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη, μεγαλύτερος βαθμό ασφάλειας. Τρίτο σημείο, διαφάνεια, πλήρης διαφάνεια. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία έτσι ώστε η δημόσια γνώμη στις χώρες μας να είναι πλήρως ενημερωμένη. Τέταρτον, θα πρέπει να ε, αναθεωρήσουμε τι τεχνικέ σε των οποίων επιλέγονται οι τοποθεσίε των ε, πυρηνικών εργοστασίων. Επόμενο σημείο, θα πρέπει να βελτιώσουμε την την ανταπόκρισή μα ε, σε ειδικέ επίγουσες καταστάσεις. Υπενθυμίζω εδώ μια πρόταση που είχαμε κάνει για μια ειδική ομάδα διάσωση. Ε, επίσης ε, θα πρέπει στην, στο κόστος να υπολογίζεται, να συνυπολογίζεται μάλλον και το κόστος της εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων είτε μέσα από ειδικέ ασφάλειε είτε με άλλους τρόπους. Ε, ε, επόμενο σημείο, ο κίνδυνος όλων των πυρηνικών ε, όλων των πυρηνικών ερευνών θα πρέπει να μελετηθεί και χαιρετίζουμε την, το σχετικό πρόγραμμα της Ευρατόμα. Επίσης θα πρέπει το, το θέμα της πυρηνικής ενέργειας να συζητηθεί από κοινού και με, την ίδια, με τον ίδιο επίγοντα χαρακτήρα που συζητούνται θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή και άλλα. Και βεβαίως ως πρώτη στο αγαθό να θεωρείται η ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες, κυρία Ούλφσκοπ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπό το φως ε, όλων όσων συνέβησαν ε, και λαμβάνοντας υπόψη και πολλές φυσικές καταστροφές ε, πέραν της Φουκουσίμα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ότι έφτασε η ώρα για μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση των, των θεμάτων και των προβλημάτων αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άμεσα να επιστήσουμε την προσοχή ε, στην καταστροφή της Φουκουσίμα. Αυτό που συνέβη την 11η Μαρτίου 2011 ήταν ε, μια καταστροφή που βεβαίως ε, ελάχιστοι ε, θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει ή φανταστεί πριν. Σεισμός και τσουνάμι που οδήγησε στο θάνατο πολλών ανθρώπων άμεσα. 340.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν και έμειναν άστεγοι. Η πόλη που βρίσκεται κοντά στην Φουκουσίμα, στα βόρεια συγκεκριμένα του πυρηνικού εργοστασίου ε, καταστράφηκε ολοσχερός ε, και ε, αυτή η περιοχή σε εύρος 25 χιλιόμετρων δεν είναι πλέον κατοικήσιμη και ξέρουμε μονάχα ότι τα σχολεία, οι άνθρωποι, η καθημερινότητα των, της, της ζωής των ανθρώπων αυτών έχουν πληγεί βαθύτατα. η Φουκουσίμα δεν υπήρξε μονάχα ανθρώπινη ή ανθρωπιστική καταστροφή. Ε, υπήρξε ένα σημείο, μια κρίσιμη καμπή στη συζήτηση για την ε, πυρηνική ενέργεια, για την δυνατότητα χρήσης δηλαδή της ενέργειας αυτής ως ε, πηγή ε, ενέργειας. Στο, τι μέλλον θα πρέπει να έχει η πυρηνική ενέργεια. έστω και αν η σχετική τεχνολογία ε, ε, προωθείται και έστω και αν οπωσδήποτε μπορεί στο εγγύς μέλλον να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ε, η πυρηνική ενέργεια και έστω και αν κάποιες χώρες ε, επιλέξουν να συνεχίζουν να οικοδομούν πυρηνικά εργοστάσια ξεκίνησε μια μεγάλη διαδικασία σκέψης όσον αφορά τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρουμε ότι η πυρηνική ενέργεια κοστίζει πάρα πολύ. Βεβαίως είναι σαφές ότι οι χώρες έχουν την δυνατότητα επιλογής, αλλά οι πολιτικές επιλογές θα πρέπει να γίνουν με τρόπο ώστε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να είμαστε σε θέση να ε, προβλέψουμε ένα ενεργειακό μέλλον που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι ε, η πρόκληση για το μέλλον. Θεωρούμε ότι δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα ε, και τουλάχιστον δεν έχει αναπτυχθεί με αποτελεσματικό τρόπο το, η εναλλακτική λύση των ε, εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα, την ανάπτυξη, τις νέες υποδομές, στο γεγονός δηλαδή ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν αυτές οι νέες πηγές ενέργειας που είναι πιο φιλικές προς την κοινωνία. Ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση αυτή και εδώ ε, κάνουμε τη συζήτηση αυτή βεβαίως με έναυσμα ε, την μνήμη των θυμάτων της Φουκουσίμα αλλά και σαν έναυσμα ε, για την μελλοντική στάση που θα έχουμε. Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους, κυρία Βαλεάν, για δύο λεπτά. Θα ήθελα εκ μέρους των ε, φιλελευθέρων να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και εγώ και την αλληλεγγύη μου για τα θύματα αυτής της καταστροφής. Θα πρέπει να προσφέρουμε την ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ιαπωνία και η περιοχή αυτή. Η πολιτική αποκρίτηση της Ευρώπης ε, σε αυτή την καταστροφή ήταν ικανοποιητική κατά τη γνώμη μας. Το σημαντικό ήταν να μην ληφθούν α, δραματικές αποφάσεις με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις υπό την πίεση της στιγμής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατάφερε να ε, συντονιστεί και να διεξάγει εθελοντικά stress test που κατά τη γνώμη μας ήταν η σωστή κίνηση. Η δική μας ομάδα αναμένει την τελική έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί το 2012 τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είμαστε πεπισμένοι πως όλα τα κατάλληλα μέτρα θα ληφθούν έτσι ώστε να εξασφαλιστούν πως τα πυρηνικά μας εργοστάσια είναι ασφαλή και μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και τρομοκρατική επίθεση. Αναγνωρίζουμε παρόλα αυτά πως είναι αδύνατο να έχουμε ένα κόσμο που θα έχει απαλλαχθεί από τον κίνδυνο 100%. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι ποιο θα είναι το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινή απάντηση και στην πραγματικότητα ε, είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους οι απόψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι σημαίνει πυρηνική ενέργεια και αν πρέπει να αποτελεί τμήμα του εθνικού ενεργειακού μείγματος. Δεν έχουμε λοιπόν μια κοινή απόκριση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στην ασφάλεια ε, των πυρηνικών εγκαταστάσεων είδατε αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία και πώς φώτισε αυτό τον κίνδυνο που ενέχουν αυτέ οι εγκαταστάσεις. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Νομίζω ότι λοιπόν θα πρέπει να πιέσουν οι κυβερνήσεις και να επενδύσουν σε ΑΠΕ έτσι ώστε να έχουμε ενέργεια η οποία θα είναι ασφαλής, θα είναι αξιόπιστη, θα είναι καθαρή και μπορεί βέβαια την πυρηνική ενέργεια για ένα χρονικό διάστημα να τη δεχτούμε ως τμήμα του ενεργειακού μας μείγματος. Νομίζω ότι θα πρέπει στο μέλλον να κάνουμε κάποιες διαφορετικές επιλογές. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Κυρία Χάμψη για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την συζήτηση αυτή, την ανασκόπηση των γεγονότων στην Ιαπωνία πριν από ένα έτος. Θεωρώ πως είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο έγινε σε πολλές χώρες το Σαββατοκυριακό το πόσο έντονο είναι το μήνυμα το οποίο στείλαμε με την Ιαπωνία πως συμμεριζόμαστε τη θλίψη ολόκληρου του Ιαπωνικού λαού. Θεωρώ όμως πως ένα χρόνο μετά από αυτή την καταστροφή πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο λεπτομερώς. Την τελευταία εβδομάδα είχα επισκέπτες από την Ιαπωνία στις Βρυξέλλες οι οποίοι, τους γνώρισα σε ταξίδι που έκανα στην Ιαπωνία επικεφαλής ήταν ο Σάκουσάτο κυβερνήτης επί 18 ετή της περιφέρειας της Φουκουσίμα ολόκληρη η αντιπροσωπεία της περιφέρειας απεύθυνε έκκληση στους Ευρωπαίους την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Οι άνθρωποι της περιφέρειας της Φουκουσίμα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση και μέχρι σήμερα αισθάνονται μόνοι. Δεν έχουν την εντύπωση πως η Ιαπωνική κυβέρνηση ασχολείται σοβαρά με την προστασία τους, μεταξύ άλλων γιατί οι οριακές τιμές για τον πληθυσμό που ζει γύρω από τη Φουκουσίμα ανέβηκαν τόσο πολύ και έφτασαν σε αυτό το οποίο ισχύει για εργαζόμενους στους πιο ε, εσωτερικούς χώρους ενός πυρηνικού εργοστασίου. Άρα πλέον σοβαρά στην Ιαπωνία συνειδητά αναλαμβάνουν τον κίνδυνο για τις επόμενες γενιές να έχουν καρκίνους και θανάτους από ραδιενέργεια. Η Ευρώπη και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θα πρέπει επιτέλους να μπορεί να αντιδρά σε τέτοιες καταστροφές. Δεν είναι δυνατόν να κλείνει τα μάτια εξαναγκαζόμενη από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στην οποία πρέπει να ασκήσει κριτική και η Ευρατόμ και τα κρατημέλη για αυτό το οποίο ισχυρίζεται πως το ε, πως Φουκουσίμα το εργοστάσιο είναι υπό έλεγχο μέχρι σήμερα δεν συμφωνούν οι Ιάπωνες ειδικοί για το ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων στα ερήπια της Φουκουσίμα. Κανείς δεν μπορεί να πει πόσα καύσιμα εξακολουθούν να ακτινοβολούν. Δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Ανα πάσα στιγμή ένας σεισμός μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των υπολείπων εκτηρίων, και να έχουμε άλλη μια καταστροφή. Η Διεθνής ε, Υπηρεσία Ατομικής ενέργειας έχει στόχο να διαδώσει την ατομική ενέργεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε σε αυτούς την ευθύνη αυτής της κατάστασης εξ ονόματος ολόκληρου του κόσμου. Οι παρακλήσεις από την Ιαπωνία των πολιτικών και των ειδικών και των αγροτών και των πολιτών είναι στείλτε μας μια διεθνή δύναμη με την εμπειρία που ε, έχει η Ευρώπη από το Τσερνομπίλ και μπορούμε έτσι να σώσουμε ζωές και ίσως να σταθεροποιηθεί η εγκατάσταση. Η σκληρότερη κριτική που ακούγεται από την Ιαπωνία είναι για τα stress test. Τώρα κάνουν και στην Ιαπωνία. Από τους 54 αντιδραστήρες αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο δύο. Οι υπόλοιποι εξετάζονται μηχανική της το ΣΥΜΠΑ. Δηλαδή μιλάμε άνθρωποι του συστήματος αυτού μου εξήγησαν πως εάν έκαναν αυτά τα stress test ένα χρόνο πριν στην ίδια τη Φουκουσίμα θα περνούσε το τεστ εξαιρετικά το εργοστάσιο αυτό. Οπότε τα stress test αυτά είναι πραγματικά αμφίβολα. Ο ισχυρισμός πως με αυτά τα τεστ ε, θα έχουμε περισσότερη ασφάλεια θα εξεταστεί στην επόμενη καταστροφή. Ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι πως ένα ε, εργοστάσιο το οποίο εμείς θα είχαμε περάσει στο τεστ αυτό στην Ευρώπη δεν θα άντεχε στην Ιαπωνία. Πρέπει να σκεφτούμε εδώ πέρα τι έχει να προσφέρει η Ευρώπη. Οι γνώσεις μας για την ενεργειακή αλλαγή και από την εμπειρία του Τσενομπίλ αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Αλλά οπωσδήποτε δεν χρειάζονται τα stress test τα ευρωπαϊκά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί έχουν το λόγο. Ο κύριος Καρύμ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα, όπως και εσείς ο ίδιος, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου ε, σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή της Ιαπωνίας πριν από ένα χρόνο. 90.000 ε, κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή και αυτή τη στιγμή ακόμα δεν θέλουν να επιστρέψουν στις πόλεις τους γιατί κατά 25 φορές ξεπερνούν οι μετρήσεις ε, της, ε, την ακτινοβολία, ε, το επιτρεπτό όριο μάλλον της ακτινοβολίας. Πριν από ένα χρόνο δημιουργήθηκε μια αμφισβήτηση γύρω από την πυρηνική ενέργεια μετά από το σεισμό και το τσουνάμι που έπληξε την Φουκουσίμα. Ε, βεβαίως ε, ύψιστη προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί για όλους μας ε, η ασφάλεια και βεβαίως θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή να οικοδομήσουμε τις νέες βάσει των βελτίστων τεχνολογικών πρακτικών θα πρέπει όλες οι μελέτες να γίνουν βάσει των σωστών ευρημάτων και των σωστών στοιχείων. Το περιστατικό της Φουκουσίμα αποδεικνύει ότι δύο φυσικές καταστροφές ωραιότητα μπορούν να συμβούν ταυτοχρόνως ε, και να ε, αντιμετωπιστούν ε, εν μέρη γιατί η Φουκουσίμα θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει το σεισμό αλλά όχι το 20 μέτρο τσουνάμι. Είναι σημαντικό να μάθουμε το μάθημα που μας έδωσε η ανταπόκριση των Ιαπώνων στην κρίση αυτή και βεβαίω θα πρέπει όλες μας οι δικλείδες ασφαλείας να μελετώνται υπό το πρίσμα του ενδεχομένου τέτοιων μεγάλων ε, κρίσεων. Ε, θα πρέπει να ε, ε, συζητηθούν από την στιγμή εξ αρχής τα προβλήματα αυτά έτσι ώστε να μην υπάρχει αποσπασματική αντιμετώπιση και διαφορετική από περίπτωση σε περίπτωση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εξεπλάγημεν όλοι θετικά από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι Ιάπωνες την κατάσταση. Η Ευρώπη τώρα από τη δικιά της μεριά θα πρέπει να μάθει το μάθημα της Φουκουσίμα και να το εφαρμόσει τα τεστ αντοχής, αυτά τα stress tests, ε, έτσι ώστε και η ασφάλεια ε, παθητική και ενεργητική να καλυφθεί ε, η έρευνα και η τεχνολογία θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού έτσι ώστε να υπάρξει η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών άμεσα. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας μας απασχολεί όλους και θα πρέπει να είναι σημαντική προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ για την ε, Νέα Ευρωπαϊκή Αριστερά, η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από ένα χρόνο αντιμετωπίσαμε ε, το φρικτό συνδυασμό σεισμού τσουνάμι και βιομηχανικού ατυχήματος και ξέρουμε όλοι ποιες ήταν οι συνέπειες. Σήμερα θέλουμε να αποτίσουμε ένα φόρο τιμή στα χιλιάδες θύματα της Φουκουσίμα και αυτό που χρειάζεται είναι να μάθουμε ποιο είναι το δίδαγμα αυτής της καταστροφής και πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές και Μιλώ για φυσικές καταστροφές γιατί τις πυρηνικές κανονικά θα έπρεπε να τι αποφεύγουμε. Δυστυχώ όμως εξακολουθούμε ένα χρόνο μετά τη Φουκουσίμα να κατασκευάζουμε νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένα χρόνο μετά τη Φουκουσίμα αυτή τη στιγμή ε, σχεδιάζονται ε, και θα οικοδομηθούν πολλές ακόμα πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η Ιαπωνία στο συλλογικό της ε, μνημονικό έχει πυρηνικές καταστροφές όπως το και τη Χειροσύμα και εμείς στην Ευρώπη έχουμε ακόμα τις συνέπειες του Τσερνομπίλ. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση η οποία δεν θα έπρεπε να έχει κλείσει. Είναι η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Πριν από πολλά χρόνια ήταν αδιαμφισβήτητη η αξία της πυρηνικής ενέργειας του για τους Ιάπωνες. Και σήμερα δύο τρίτα της χώρας την απορρίπτουν γιατί γνωρίζουν πως ε, ο αριθμός θυμάτων είναι τέτοιος σε μια ενδεχόμενη καταστροφή που πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο. Είναι οι πολλές γενιές που χάθηκαν και η πολιτική ε, η δική μας, η άτολμη, ε, είναι μια πολιτική η οποία δείχνει μια υπεροψία ε, των κρατών, μια και οι πολίτες στην Ευρώπη ζητούν να μην χρησιμοποιούμε πυρηνική ενέργεια και παρόλα αυτά οι κυβερνητικές επιλογές δεν αλλάζουν. 300.000 εκτοπισμένοι στην Ιαπωνία, 100.000 εκ των οποίων δεν θα γυρίσουν ποτέ σπίτι τους. Και αυτό το οποίο στο παρελθόν ήταν η ο δικός τους χώρος είναι πια ερήπια, ε, κατεστραμμένα σπίτια, ε, ραδιενέργεια, ε, απειλή, ε, ραδιενεργά ύδατα, εδάφη. Δεν μπορεί καν να πάει κανείς να επισκεφτεί αυτά τα ερήπια, όπως πηγαίνει και επισκέπτεται τα ρωμαϊκά ερήπια, τα ερήπια των Μάγια. Παρ' όλα αυτά, η Φουκουσίμα ε, είναι τα ερήπια ενός πολιτισμού και τα ερήπια της Φουκουσίμα είναι τα ερήπια ενός πολιτισμού που αποφάσισε στον αναπτυξιακό της μοντέλο να ε, εντάξει αυτή τη θανατηφόρο τεχνολογία. Δεν φταίει ούτε ο σεισμός ούτε το τσουνάμι. Η πυρηνική όμως καταστροφή ε, έχει ενόχους που την προκάλεσαν. Στην Ιαπωνία όπως και στην Ευρώπη έχουν κινητοποιηθεί οι πολίτες κατά της πυρηνικής ενέργειας γιατί γνωρίζουν στην Ιαπωνία πως δεν υπάρχει σίγουρη πυρηνική τεχνολογία. Ξέρουν πως δεν υπάρχει καμία μια δυνατότητα ε, να αντέξει και δεν υπάρχουν και τρεις, τρεις τεστ που να ομοιάζουν ε, στα όσα συνέβησαν και χτύπησαν τη Φουκουσίμα. Εντάξει, είναι εθνική επιλογή και εθνική αρμοδιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να έχουμε σύνορα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σπερόνι θα ήθελε το λόγο για δύο λεπτά για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τραγωδία της Φουκουσίμα κατέδειξε μετά το Τσερνομπίλ ότι δεν υφίσταται ακόμα η πλήρης ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είναι γεγονός ότι οι δύο περιπτώσεις διαφέρουν. Στην περίπτωση του Τσερνομπίλ ε, υπήρξε εσωτερικό πρόβλημα ε, στον αντιδραστήρα, ενώ για την περίπτωση της Φουκουσίμα τα αίτια ήταν εξωτερικά, δηλαδή ε, ένας σεισμός και ένα παλιροϊκό κύμα τρομερής έντασης και ύψους πρωτογνώριστο στην ιστορία του πλανήτη. Βεβαίως με όλες αυτές τις περιπτώσεις και τα περιστατικά αρχίζουμε να σκεφτόμαστε περισσότερο το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Πολλοί μας λένε ότι θα πρέπει να ε, σταματήσουμε τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, έστω και αν πολλές χώρες εξαρτώνται από αυτήν. Είναι γεγονός ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει μία σε βάθος συζήτηση και σκέψη ε, για το θέμα αυτό. Και βεβαίως έχει αντιληφθεί και ορθώς ότι είναι εθνική διαδικασία και αρμοδιότητα το θέμα της πυρηνικής ενέργειας αλλά και εμείς εδώ θα πρέπει να έχουμε λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σκεφτόμαστε βεβαίως όλα τα θύματα της, της τραγωδίας. Ευχαριστώ. Κύριε Σφερώνη, η κυρία Ρέντινγκ τώρα για την Κομισιόν. Κύριε Ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνος πέρασε από την τρομακτική καταστροφή, την πυρηνική καταστροφή στην Ιαπωνία. Ένα από τα χειρότερα ατυχήματα που έχουν γραφτεί στην ιστορία της ειρηνική πυρηνικής τεχνολογίας. Είμαστε λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή εδώ για να δούμε ποια είναι τα διδάγματα τα οποία μάθαμε από το τη Φουκουσίμα αλλά και για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στον Ιαπωνικό λαό πριν τη Φουκουσίμα, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροφή είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια βελτίωσης πυρηνική ασφάλειας, έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση που θα βασίζεται σε εχέγγυα ασφάλειας, υψηλά πρότυπα και έχουμε βέβαια και την οδηγία του 2009, όπως επίσης και μετά την οδηγία του 2011 για την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον επικοδομητικό του ρόλο στην έγκριση αυτών των δύο κομβικών οδηγίων. Μετά το ατύχημα στην Φουκουσίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια σφαιρική και πλήρη αξιολόγηση όλων των πυρηνικών σταθμών που λειτουργούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως επίσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε πως αυτά τα stress test έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2011 και βασίζονται σε μια κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία και πρέπει να σας πω ότι άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα είπε η κυρία Χάρμς και θα σας πω ότι θα μεταφέρω ε, τα σχόλιά σας στον Επίτροπο Ότιγκερ. Όλα τα κράτη-μέλη που έχουν πυρηνικούς σταθμούς και η Λιθουανία η οποία αποξυλώνει τις μονάδες που παράγουν πυρηνική ενέργεια συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική αξιολόγηση και έχουν υποβάλει εθνικές εκθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή αναθεωρούνται από τους ομολόγους τους. Ε, ξέρετε και πως οι γειτονικές μας χώρες έχουν ε, συστρατευτεί και αυτές με την μεθοδολογία μας και συμμετέχουν η Ελβετία και η Ουκρανία στην αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα αυτών των peer review που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της διαδικασίας θα δοθούν ε, στη δημοσιότητα μέχρι τέλη Απριλίου και η τελική μας έκθεση θα παρουσιαστεί ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον συνάδελφο Ότιγκερ τέλη Ιουνίου του 2012 μου ζήτησε να σας μεταφέρω πως θα είναι διαθέσιμος και για την συζήτηση του θέματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όποτε χρειαστεί τα συμπεράσματα από αυτά τα stress test θεωρούμε πως θα αποτελέσουν μια αντικειμενική αξιολόγηση της ποινική ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσουν και τη βάση για νομοθετικές ή μη νομοθετικές προτάσεις που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθούν οι επιδόσεις μας ε, στην ενέργεια. Βασική κλάδη είναι οι τεχνικές απαιτήσει για την ασφάλεια, η διαχείριση και βεβαίως η η απόκριση αλλά και τα επίπεδα ετοιμότητας. Έχουμε και κάποιες απειλές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ε, κακόβουλες ε, επιθέσεις λαμβάνονται υπόψη και έχουμε μια ομάδα ad hoc για την πυρηνική ασφάλεια που στο, Ευρω... στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητά το θέμα αυτό και τα πρώτα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε μια τελική έκθεση τον Ιούνιο. Η έκθεση αυτή θα επισυναυθεί στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποβληθεί προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και προς το Κοινοβούλιο. Ξέρετε πως η εφαρμογή των ε, συστάσεων που θα προκύψουν αποτελούν εθνική αρμοδιότητα. Όμως, η επιτήρηση και οι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων πεπραγμένων θα πρέπει να εξασφαλίσουν πως εφαρμόζονται οι απαραίτητες βελτιώσεις για την ασφάλεια και τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν έτσι ώστε τα κατάλληλα μέτρα να ληφθούν για να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα επίπεδα ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει δραστήρια όλες τις εξελίξεις και τέλος αλλά όχι ως σημασίας, θα πρέπει να έχουμε μια κουλτούρα ασφάλειας και θα πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Γιατί? Γιατί αυτά τα stress test αποτελούν ένα σημείο αναφορά σε διεθνή επίπεδο, ένα benchmark. Και από την πρώτη στιγμή εμεί εμπλέξαμε στη διαδικασία τι γειτονικέ μα χώρε για να μην είμαστε οι μόνοι που θα κάνουμε κάτι παρόμοιο, αλλά για να επεκτείνουμε αυτή την ε, κουλτούρα ασφάλειας και στα σύνορά μας. Διεθνή συνεργασία λοιπόν, κυρίως στα πλαίσια της ε, Διεθνής Υπηρεσίας Ενέργειας. Εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικό να συνεργαζόμαστε και έχουμε σκοπό να συνεισφέρουμε στην ενημέρωση της Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, να είναι καλύτερη, πιο εύκολα διαχειρίσιμη και βεβαίως να επιβάλλεται καλύτερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε και το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την ισότητα των φύλων. Και επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να πω ότι αποτελεί έτσι κι αλλιώ